Αυτά ήθελα να πω. Να ευχαριστήσω όλους όσους ε, μίλησαν υπέρ τη εκθέσεω μου ε, και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς για την εργασία που κάνατε ως ε, εισηγήτρια και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει το ζήτημα. Λοιπόν, θα, στα, θα ε, ληφθούν οι τελικές αποφάσεις μέσω της ψηφοφορίας στις 12.30 αύριο. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση του κυρίου Κρόιτσμαν. Τελωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία. Αυτός είναι ο τίτλος της εκθέσεως. Ο εισηγητή έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, Κύριε... Πρόεδρε κύριε κυρίες και κύριοι, η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει υπαρξιακή σημασία για την ευρωπαϊκή επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. Έχουμε διαρκώς προβλήματα παραβίασης που απειλούν την ανάπτυξη των οικονομιών μας και η απομίμηση προϊόντων όχι μόνο βλάπτει τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις αλλά μπορεί να είναι και κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια την ίδια την ευζοία των, καταναλωτών μας. Οι τελωνιακές αρχές στα εξωτερικά σύνορα βρίσκονται σε μια σχετικά ευνοϊκή θέση να μπορούν να αναχαιτήσουν τις ροές αυτών των προϊόντων απομίμησης προτού φτάσουν στις αγορές μας. Γι' αυτό θα πρέπει να προσαρμοστούν οι διατάξεις στις ανάγκες. Αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την ανάγκη και πέρσι υπέβαλε μια καλή πρόταση διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής ασφαλίζοντας ένα υψηλότερο επίπεδο ε, αντιμετώπισης προϊόντων απομίμησης, προϊόντων μαϊμούδων, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα σημαντικό δυναμικό ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί θα πρέπει οι τελωνιακές αρχές ε, να μπορούν να δράσουν ακόμα πιο αποτελεσματικά. Στην έκθεσή μου έχω κάποιους κύριους άξονες που παρακολουθώ. Προστασία της, ε, ε, ενίσχυσης της προστασίας των καταναλωτών, ενίσχυση της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, προστασία των καταναλωτών. Αντίθετα με κάποια άποψη η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κυρίως προς όφελος των καταναλωτών διότι τα προϊόντα απομίμησης ε, και, παρα, ε, και παράτυπα προϊόντα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις ε, προδιαγραφές ασφάλειας ούτε στην ανάγκη προστασίας της υγείας των καταναλωτών. Έχουμε ανησυχητικές εικόνες και γεγονότα μέσω προϊόντων μαϊμούδων για την ίδια την υγεία των καταναλωτών ένας ε, Γερμανός ε, ε, βιομήχανος, αυτοκινητοβιομήχανος μου επεσήμανε πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος παραποιημένων συστημάτων για τα φρένα των αυτοκινήτων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά με τα προϊόντα μαϊμούδες. Έχουμε κάνει κάθε προσπάθεια να διευκολυνθεί το έργο των τελωνιακών αρχών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ή δυνατόν ενιαίο πλαίσιο ανείχνευσης και καταστροφής προϊόντων προϊόντων απομίμησης ε, από τις τελωνιακές ε, αρχές. Η δική μας ε, πρόταση χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανάμειξη τρίτου δίνει τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να καταστρέφουν αυτά τα αντικείμενα. Έτσι η προστασία, η νομική προστασία μέσα στο πλαίσιο κράτους δικαίου διασφαλίζεται. Η ειδική αντιμετώπιση των μικρών αποστολών διευκολύνει τις τελωνιακές αρχές, διότι δεν τις επιβαρύνει. Έτσι και οι τελωνιακές αρχές και οι χρήστες εποφελούνται και η ανταλλαγή στοιχείων σε σχέση με τις αρμόδιες τελωνιακές αρχές τρίτων χωρών θα πρέπει να βελτιώνεται για την ε, διακίνηση των προϊόντων αυτών που πρέπει να καταπολεμηθεί στην ίδια την πηγή και ιδιαίτερα η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που πρέπει να διασφαλίζεται. Διότι αυτή η πνευματική ιδιοκτησία είναι που δημιουργεί καινοτομία στην Ευρώπη και θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία στην Ευρώπη προστατεύοντας τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών. Υποβάλουμε προτάσεις ε, ώστε να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε σχέση με την ε, μοίρα των προϊόντων αυτών η πνευματική ιδιοκτήτη του αρχικού προϊόντος. Θα πρέπει μέσα στο πλαίσιο των ε, εξοδικαστικών διαδικασιών να λαμβάνονται αυτά υπόψη. Τρίτον, η μεγαλύτερη βελτίωση είναι η ανατροπή του βάρους αποδείξεως. Στη συνέχεια θα επισέλθω περισσότερο σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Σέμετα και να του ζητήσω να λάβει εκείνο τον λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Ε, χαίρομαι για την συμφωνία των αρμοδίων επιτροπών στην πρότασή μας. Ο κύριος Κρόισμαν έκανε εξαιρετική δουλειά στην έκθεση αυτή και είναι επιταγή να ε, προστατεύουμε τα ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη και πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι θα εφαρμόζονται διότι θα ήθελα σχολιάζοντας να αναφέρω τρία μηνύματα. Καταρχήν ότι ε, το μόνο δικαίωμα δίδεται μέσω της εφαρμογής. Ε, τα, ε, θα πρέπει δηλαδή και τα τελωνία να επιβάλλει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Εάν υπάρχουν παραδιευιάσεις δεν θα πρέπει να ξεφεύγουν από ότι κανονισμό και αν ε, ε, δεν ε, υπάρχει εφαρμογή σε περίπτωση που δεν υπάρχει δικαίωμα τι γίνεται κατά τη διέλευση των συνόρων χωρίς να έχει συζητηθεί η αρμοδιότητα των αρμοδίων αρχών διότι δεν βλέπουμε εις τις ε, το δίκαιο να υπάρχει μία πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αυτές οπότε ε, θα πρέπει ε, σε περίπτωση παραβιάσεων ε, οι πέτοι να φεθούν ελεύθεροι διότι δεν υπάρχει απόδειξη παραβίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω βεβαίως το πρόβλημα που υπάρχει με τα φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο επιλύσαμε με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων των διεθνών ομολόγων μας και αλλάζοντας και ε, ε, τροποποιώντας την νομοθεσία. Ε, γι' αυτό και χαιρετίζω την τροπολογία που κατετέθη την τελευταία στιγμή σχετικά με την παρακολούθηση. Όσον αφορά την καταστροφή των προϊόντων σε περίπτωση παραβιάσεως των διπλωμάτων πνευματικής ιδιοτεξίας, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να υπάρξει χωρίς να υπάρχει ρητή συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων. Θα χρειαστεί δηλαδή να έχουμε μία πρακτική και λογική προσέγγιση και ε, εάν υπάρχουν μικρές αποστολές θα πρέπει να έχουμε το σωστό ορισμό που να μπορεί να εφαρμόζεται στην πρακτική. Ε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε νέες κατευθύνσεις ε, και να υπάρξουν κατεξουσιοδότης πράξεις οι οποίες θα ρυθμίσουν τα θέματα αυτά. Διότι μπορεί κανείς να επέμβει μόνο όταν υπάρχουν σωστές αποδείξεις και θα πρέπει ε, τα ε, τελωνία να αιτιολογούν ε, γιατί θέλουν να κατακρατήσουν τα εμπορεύματα. Ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει μία σωστή εφαρμογή της των αρχών της πνευματικής ιδιοκτησίας και αυτό να αποτελέσει τον χρυσού κανόνα σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ εν ονόματι της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ η κυρία Μπαντία Ικουτσέτ. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, Παγκοσμίου Εμπορίου θα ήθελα να τονίσω πρώτα απ' όλα τη σημασία αυτού του κανονισμού και για το εμπόριο και για τους καταναλωτές. Μια και θέλει να ενισχύσει τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση προϊόντων απομίμησης και μαϊμούδων που έχει τόσο αυξηθεί και είναι τόσο ανησυχητικό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ρόλο των τελωνιακών αρχών για την προστασία των πνευματικών αυτών των δικαιωμάτων χωρίς αλλαγή του νομικού πλαισίου. Μια μεταρρύθμιση λοιπόν αυτού του νομικού πλαισίου είναι απόλυτα αναγκαία και σε ένα προσεχώς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη αυτές τις ανάγκες και θα καλύπτουν τις ανάγκες προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Και για τα γενώσιμα φάρμακα τα οποία βρίσκονται υπό διαμετακόμιση για να αποφύγουμε να ε, ε τροχοπεδούνται, να σταματούν στα σύνορα θα πρέπει να Εντάξει, να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκε τρίτων χωρών που τα χρειάζονται για χρήση τους. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε. Εξ του ΕΛΚ, η κυρία Γκάλιο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του κανονισμού 2003 συμπίπτει με μια γενικότερη συνειδητοποίηση των ζημιών που προκύπτουν από την παραχάραξη και όσον αφορά την ασφάλεια αλλά και την υγεία των ε, πολιτών της Ευρώπης ε, που απειλείται γιατί βεβαίως η παραχάραξη αφορά ε, και τα παιδικά παιχνίδια αλλά και προϊόντα υγιεινής και φάρμακα. 250 ε, δις από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κάθε χρόνο λόγω της παραχάραξης ε, που ε, κάθε χρόνο επίσης καταδικάζει σε ανεργία 100.000 εργαζόμενους χάνονται οι αντίστοιχε θέσει εργασία δηλαδή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Κρόιτσμαν γιατί η Επιτροπή ΙΝΚΟ δούλεψε με μεγάλη ευφυΐα ε, και με πολύ ορθό τρόπο ε, έτσι ώστε να φτάσει σε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα το οποίο και προστατεύει τους έχοντες δίκαιο αλλά ε, και προτείνει και εναλλακτικέ λύσεις. Βεβαίως τα, οι παράλληλες εισαγωγές και τα προσωπικά, ε, οι προσωπικές αποσκευές έχουν ε, ε, βγει έξω από, την, από το πεδίο. Ο καταναλωτής, ο τελικός καταναλωτής θα είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να προστατευτεί. Όσον αφορά τώρα τα γενώσιμα φάρμακα, εδώ έχουμε αποσαφηνίσει το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να ταυτιστεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Οι σοσιαλιστές και οι Γκουε ζήτησαν πιο αυστηρό έλεγχο μέσω τροπολογιών ε, το, της παρέμβασης των τελωνιακών αργών και το ΕΛΚ θα στηρίξει τις τροπολογίες αυτές 109, 110 και 121. Τέλος, ε, στο Συμβούλιο έχει προταθεί συμβιβαστικό κείμενο από την Προεδρία και έχει γίνει δεχτή ε, ε, τη 14η Ιουνίου 2012 και επομένως θα ολοκληρωθεί η θέση του Κοινοβουλίου έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η κυρία Χέτ. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω την αναδιατύπωση, την αναθεώρηση του κανονισμού και ευχαριστώ τον κύριο Κρόισμαν για την πολύ θετική συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές. Πολλά αγαθά έχουν ενταχθεί και είναι άμεσα ε, για υπέρ των καταναλωτών. Παιχνίδια, φάρμακα, που μπορούν να οδηγήσουν σε οποιασδήποτε βλαπτικές επιπτώσεις για την υγεία. Γι' αυτό πρέπει να προσφέρουμε ασφάλεια στην ενιαία εσωτερική αγορά. Αυτό είναι υποφελέ για τους καταναλωτές. Και γι' αυτόν τον λόγο αγαθά που εισάγονται για ιδιωτική χρήση ή παράλληλες εισαγωγές πρέπει να την χάνουν εξαίρεσης. Στην Επιτροπή ΙΜΚΟ αυτό που θέλουμε είναι και τα εμπορεύματα, τα αγαθά υποδιαμετακόμιση να λαμβάνονται υπόψη και να καλύπτονται. Όμως εδώ πρόσθετα στοιχεία είναι αναγκαία για την πρόσβαση στα γενώσιμα φάρμακα που μπορεί να δυσχερανθεί η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα στα γενώσιμα μέσω αυτών των διαδικασιών. Γι' αυτό με την Νομική Επιτροπή ε, έχουμε προετοιμάσει κάποιες ε, ε ώστε η πρόσβαση στα γενώσιμα να διασφαλίζεται παρόλα αυτά. Η κυριότερη τροπολογία Βιβλία αναφέρεται στο ότι τα αγαθά θα πρέπει να αποκλείονται. Να αποκλείονται αγαθά εκτός αν υπάρχουν επαρκή τεκμήρια και στοιχεία ότι πρόκειται για αγαθά τα οποία θα εισάγονται ή θα χρησιμοποιηθούν στις ευρωπαϊκές αγορές και για τα γενώσιμα θα υπερψηφίσουμε το κείμενο του κυρίου Κρόιτσμαν. Είναι μια προστευμένη διαδικασία, δεν θα πρέπει όμως να ισχύει για άλλου είδους αγαθά, <clears throat> για προϊόντα πειρατείας ε, ή απομίμησης ή προϊόντα μαϊμούδες διότι διαφορετικά θα υπάρξουν μεγάλες δυσκολίες στη διαμετακόμιση για τα γενώσιμα. Η ΙΝΚΟ τοποθετήθηκε από αυτού του θέματος και έτσι υπάρχει μπορώ να πω ένας ε, κίνδυνος να κατασχεθούν γενώσιμα φάρμακα και η διασυνοριακή ε, κυκλοφορία διακίνηση αυτών των φαρμάκων να δυσχερανθεί. Χρειαζόμαστε νόμιμα γενώσιμα φάρμακα. Είναι υπέρ των συμφερόντων των καταναλωτών. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούν οι σοσιαλιστές να δυσχεραίνεται η πρόσβαση στα γενώσιμα, ενώ τα χρειάζονται για την ευζοία και την υγεία τους οι καταναλωτές. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Μάντερς θα ελάμβανε τον λόγο εξ ονόματος φιλελευθέρων αλλά δεν παρίσταται από ό,τι μπορώ να διαπιστώσω. Γι' αυτό ο κύριος Έγκστρομ θα έχει τώρα την ευκαιρία να παρέμβει και να μας γνωστοποιήσει τις απόψεις του εξ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε όλοι ότι τα παραποιημένα προϊόντα είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θυμίσω όμως τους συναδέλφους ότι ήδη υπάρχει πολλή νομοθεσία όσον αφορά τα θέματα αυτά. Το νέο σε αυτή την έκθεση είναι ότι επεκτείνει την ευθύνη των τελωνίων ε, στην δυνατότητά τους να σταματούν τα παραποιημένα προϊόντα ε, και ε, να ασχοληθεί πλέον το τελωνίο με κάθε είδους επιβολή για όλα τα δικαιώματα διανοητικής η ιδιοκτησία. Πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι εξαιρετικά περίπλοκα και πολύ εξειδικευμένα και επομένως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει ο απλός τελωνιακός υπάλληλο έτσι και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία. Ε, όσον αφορά την πρόσβαση στα, όσον αφορά τα γενώσιμα φάρμακα, οι οργανισμοί οι οποίοι δουλεύουν ε, ακριβώς έχοντα θέμα την πρόσβαση στα φάρμακα δουλεύουν πάρα πολύ και για τα θέματα αυτό ε, και ε, συμφωνούμε ότι εδώ μπορεί να υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα. Εγώ θα ήθελα όμω να θίξω και κάτι άλλο. Ε, νομίζω ότι αυτή η εστίαση που έχουμε ε, σε μικρά πράγματα μερικές φορές ε, μπορεί να μας οδηγεί σε προβλήματα. Ε, ένας απλός ε, ε, πολίτης ο οποίος περνάει από το τελωνίο και βλέπει ότι του κατάσχουν το smartphone του γιατί υποτίθεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μα αυτός ο άνθρωπος θα χάσει τελικά την εμπιστοσύνη που έχει στα τελωνία θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πολύ Ανδρέας Βάμπ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Κρόισμαν δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία διότι τα βασικά θέματα που είναι μέρος μιας στρατηγικής για την πνευματική ιδιωτικησία για ολόκληρη την Ευρώπη ένα σωστό σημείο ενάρξεως όπως άλλωστε έχει αναφερθεί. Αν θέλουμε να υπάρξουν βελτιώσεις στη διεθνές εμπόριο χρειάζεται να υπάρξουν αλλαγές οι οποίες όμως συγχρόνως θα είναι προς όφελος και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι κάθε χρόνο λόγω των παραποιήσεων έχουμε ε, ζημία 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το θέμα όσο όχι μόνο σχετικά με την εφαρμογή Τη της στρατηγικής πνευματικής ιδιοκτησίας είναι κάτι το οποίο έχω ήδη πει αλλά και από την άλλη πλευρά πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε οι νέοι να κατανοήσουν καλύτερα ότι η πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό αλλά είναι κάτι το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο επί πάρα πολύ καιρό και ως εκ τούτου κύριε Επίτροπε ε, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ πολύ θετικό ότι ο Επίτροπος μπανιέ ε, κατήρτισε αυτό το βραβείο για την πνευματική ιδιοκτησία το οποίο επιδώσαμε πέρυσι για πρώτη φορά. Η εμπλοκή των τελωνιακών αρχών στη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πειρατη... πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύει από την πειρατεία διότι ε, βεβαίως τα διπλώματα δικαιώματα βραστεχνίας πρέπει να προστατεύονται πέραν αυτού όμως και τα προϊόντα μαϊμούδες που οδηγούν σε διενέξεις σχετικά με τα διπλώματα είναι πολύ σοβαρό θέμα και γι' αυτό είναι ίσως μια πτυχή που πρέπει να ξανασυζητήσουμε με το Συμβούλιο στη δεύτερη ανάγνωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Γκέπχα τώρα. Η κυρία Γκέπχαρτ, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Κρόσμα. θα έλεγα ότι έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα ενώπιον μας που πρέπει να απαντήσουμε και να ρυθμίσουμε. Και γι' αυτό το χαιρέτησα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την νομοθετική πρόταση από πλευρά τη. Πρόκειται εδώ για την ίδια την ασφάλεια των πολιτών μας, γυναικών και ανδρών. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες που λάβαμε πόσο προβληματικά είναι αυτά τα προϊόντα μαϊμούδες και για την υγεία και για την ίδια την ευζοία και την ευημερία των πολιτών αλλά και για την ίδια την διαμόρφωση των τιμών αυτών των προϊόντων και για τους επιχειρηματίες, γυναίκες και άνδρες διότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να πολλούνται με μια τιμή που θα καλύπτει και τα θέματα της προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας που θα διασφαλίζει. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία όμως ε, με αφήσιμο τρόπο επίμαχα συζητούνται στην Ευρωβουλή. Κάποια φαίνεται ότι έχουν ρυθμιστεί. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την συνάδελφο κυρία Χέντ που έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα γενώσιμα φάρμακα. Τα φάρμακα ιδιαίτερα υποδιαμετακόμιση ως αγαθά. Είναι ένα θέμα υπαρξιακό. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να δυσχερανθεί η διακίνηση αυτών των προϊόντων που δεν έχει καμιά σχέση αυτή η επιβάρηση με την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει ιδιαίτερα προσεκτικά να σταθμίσουμε το τι κάνουμε σε σχέση με τα γενώσιμα. Κατά τα άλλα, πολύ καλά ε, καταδείχθηκαν ποια προβλήματα υπάρχουν και αντιμετωπίζουμε. Το δεύτερο σημείο το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι και το βρίσκω πολύ καλό αυτό το οποίο είπατε είπατε πιο πριν κύριε Σέμετα, Επίτροπε, για την παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και για την διασφάλιση του νομικού πλαισίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και γι' αυτό η ομάδα μας σε σχέση με τις τροπολογίες θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές για να υπάρχει νομική ασφάλεια και να υπάρχει και το κράτος δικαίου που θα διασφαλίζεται, ένα νομικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών μας ως καταναλωτών. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου αδιάφορο επιτείνω θα ψηφίσουμε στο τέλος τέλος. Γι' αυτό η τελική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο είναι κάτι ανοιχτό ακόμα ως θέμα και θα το αποφασίσουμε αύριο πώς θα ψηφίσουμε. Θα σε ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Μπάστος παρακαλώ έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την ε, τον συνάδελφο εισηγητή για, αυτό, για την έκθεση. Είναι ένα θέμα που έχει τεράστια σημασία για την Ευρώπη. Αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή οικονομική, χρηματοοικονομική κρίση και για τα κοινωνικά δικαιώματα και για τα δικαιώματα προστασία ε, τη πνευματική ιδιοκτησία, που είναι τεράστια σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ενισχύει την ανάπτυξη τη έρευνα και τη καινοτομία. Πρέπει να διασφαλίζει την επιστημονική γνώση και την τεχνολογία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Όλα αυτά προς το στόχο της δημιουργίας ανάπτυξης και δημιουργίας αναβαθμισμένων θέσεων απασχόλησης. Δυστυχώς όμως βλέπουμε σημαντική παραβίαση των δικαιωμάτων όσον αφορά τα προϊόντα μαϊμούδες με τεράστιες απώλειες. Απώλειες 250 δισεκατομμυρίων ευρώ ετήσια εις βάρος της ευρωπαϊκής και εις βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων με αυτά τα αρνητικά ε, συνεπαγόμενα για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτελούν σημαντική απειλή για την υγεία και την ευζοία και ευημερία των Ευρωπαίων καταναλωτών. Αυτά τα προϊόντα μαϊμούδες, ιδιαίτερα όταν έχουμε τρόφιμα ή φάρμακα, ή ιδιαίτερα όταν δεν, δεν σέβονται τις διατάξεις για το περιβάλλον. Γι' αυτό οι τελωνιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά αυτών των προϊόντων μαϊμούδων. Πρέπει να ενισχύσουμε τους ελέγχους σε σχέση με την ε, νομοθεσία που ισχύει, να προστατεύσουμε την Ευρώπη, να υπάρξει αποσαφήνιση της νομικής θέσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τις νέες εξελίξεις και να συνεισφέρουμε με αυτόν τον τρόπο με την καλή, για την καλύτερη προστασία της οικονομίας και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Τα πνευματικά δικαιώματα λοιπόν έχουν ιδιαίτερη προτεραιότητα και σπουδαιότητα για να προωθήσουμε τη στρατηγική του 2020 από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και τώρα ένα λεπτό αυτό. Η κυρία Ράπτη, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα που συζητάμε σήμερα έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η εμπορική και η οικονομική διάσταση. Η άλλη διάσταση είναι ηθική. Η παραποίηση των προϊόντων στοιχίζει στην οικονομία, στοιχίζει σε θέσεις εργασίας, αλλά στοιχίζει και στην ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών. Αυτή την διτή διάσταση του θέματος που συζητάμε σήμερα δεν πρέπει να την ξεχνάμε. βάζουμε λοιπόν τα τελωνία και τους τελωνειακούς υπαλλήλους ουσιαστικά να πάρουν αποφάσεις ουσίας. νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή διότι θα πρέπει μεν να υπάρχουν έλεγχοι να είναι σύμφωνα με το γράμμα του νόμου αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να υπάρχει και ευελιξία το χαρακτηριστικό παράδειγμα που απαιτεί ευελιξία είναι τα γενώσιμα φάρμακα και για να μην μασάμε τα λόγια μας και να λέμε τα πράγματα όπως είναι θέλω πραγματικά να τονίσω ότι με το πρόσχημα των παραποιημένων προϊόντων μεγάλες εταιρείες βρίσκουν ένα τρόπο βρίσκουν την ευκαιρία βρίσκουν το παραθυράκι να σταματούν γενώσιμα φάρμακα που προορίζονται για χώρες της αφρικής. πρέπει να το δούμε πραγματικά με πολύ προσοχή. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κύριε Σκοφεράτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπή, ο στόχος μας είναι να εγγυηθούμε ε, την ασφάλεια των ε, καταναλωτών ε, και βεβαίως θα πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην τους κάνουμε περισσότερο κακό κρυβόμενοι πίσω από υποτίθεται μεγαλύτερη αυστηρότητα. Ε, οι τελωνιακοί υπάλληλοι δεν έχουν ε, την ε, επαγγελματική κατάρτιση και προετοιμασία έτσι ώστε να ασχοληθούν με αυτήν την επιβολή. Κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ στα γενώσιμα φάρμακα Όμω. Τα γενώσιμα φάρμακα δεν είναι παραχαραγμένα φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν μονάχα την ενεργή, τη δραστική ουσία του προϊόντος και βεβαίω κοστίζουν πολύ λιγότερο από τα άλλα φάρμακα. Εάν δεν αποσαφινιστεί η διαφορά ανάμεσα ανάμεσα σε ένα φάρμακο ε, ειδικό και ένα φάρμακο γενώσιμο ε, θα υπάρξει μεγάλο πρόσκομα στην ε, κυκλοφορία των γενώσιμων φαρμάκων και αυτό τελικά θα αποβεί σε ζημία των καταναλωτών. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ζητούμε και σαν ομάδα τροποποίηση του κανονισμού. Κατά αυτή την έννοια ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής η κυρία Τρικογέννη Περές. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να πω, όπως και οι προλαλήσαντες, ο κύριος ε, Κοφεράτη ακριβώς, η προστασία των καταναλωτών περνάει από την ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως των σημάτων και των δικαιωμάτων δημιουργών. Και στα τελωνία πολλές φορές τα προϊόντα μαϊμούδες πάγονη κίνδυνο για την ίδια τη ζωή των καταναλωτών. Γι' αυτό πρέπει να εξοπλίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αναγκαία μέσα ώστε να αποφεύγουμε την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέτοιου είδους προϊόντων και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά έχει προτεραιότητα να υπάρξει ισορροπία μεταξύ προστασίας αποτελεσματικής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και μιας αποτελεσματικής νομοθεσίας. Να μην πέσουμε στον πειρασμό του να έχουμε μια νομοθεσία που δεν θα βασίζεται σε τεκμήρια που θα αναφέρονται σε νομικές ε, υποχρεώσεις και διατάξεις. Διότι βλέπουμε ότι έχουμε νόμιμα φάρμακα υποδιαμετακόμιση, γενώσιμα φάρμακα, τα οποία στοχεύουν σε άλλες τρίτες χώρες που τα χρειάζονται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και στη συνέχεια. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρέμβω σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, λέγει ο κύριος Κέλλη. Και θα ήθελα να επενέσω τον Επίτροπο και τον εισηγητή για τις ε, συστάσεις ε, που έγιναν, που έκαναν ιδιαίτερα όσον αφορά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι η ζημιά από τα προϊόντα μαϊμούδες ε, που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τεράστια επίπτωση. Και έχουμε και την απώλεια θέσεων απασχόλησης και τον κίνδυνο στην ίδια την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας. Είναι σαφέστατο λοιπόν ότι έχουμε ένα μείζον πρόβλημα ενώπιον μας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και ιδιαίτερα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό σε σχέση με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική οικονομική κρίση και τις τεράστιες οικονομικές απώλειες που συνεπάγονται αυτά τα προϊόντα πρέπει να κάνουμε κάτι το σημαντικό προς όφελος των πολιτών μας και προς όφελος της οικονομίας μας, ε, οικονομίας μας που πρέπει να προστατεύσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτό το φαινόμενο και να σημειωθεί πρόοδος. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. στη συνέχεια παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι. Νομίζω ότι ε, πρέπει να ανησυχούμε ε, διότι θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από προϊόντα ε, παραποιημένα που διακινούνται μέσω των συνόρων. Υπάρχουν συνεχείς απώλειες οι οποίες δεν επιτρέπουν να εφαρμόζεται είναι διασυνοριακά ε, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για να μπορέσουμε λοιπόν να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και τις νόμιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουμε μία νέα προσέγγιση στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και να μπορέσουμε ε, να εξαιρέσουμε ε, ορισμένα σημεία από αυτή την πρόταση εγώ έχω διάφορες επιφυλάξεις σχετικά με την προσέγγιση που έχει επιλεγεί για τη μεταφορά αγαθών και δεν αναφέρθηκα καν στα φάρμακα. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μέλτσε. Αυτό που για τους μεν είναι καλό, για τους άλλους είναι κακό. Αυτό γίνεται και με τα νόμιμα προϊόντα όταν υπάρχουν αντίγραφα και προχωρούν. Οι παραποιητές άλλωστε ε, κάνουν οικονομίες και στην ποιότητα των προϊόντων και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αν δούμε ε, στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι υπάρχουν κινέζικα παραποιημένα προϊόντα ε, ε, καχέκτυπα ευρωπαϊκών και είναι πολύ βασικό να μπορέσουμε να αποφύγουμε την πειρατεία χωρίς όμως να επιβαρύνουμε τους καταναλωτές διότι 85% των ε, εισαγωγών των πειρατικών προϊόντων έρχονται από την Κίνα άρα μπορούμε να ενισχύσουμε τους ελέγχους. Ευχαριστώ κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησία είναι ένα από τα κύρια οχήματα της καινοτομία και οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών ισούται με κλοπή και θα πρέπει να υφίσταται κυρώσεις. Ε, η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά και την προστασία νέων ιδεών. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και επομένως η πειρατεία και η παραχάραξη των προϊόντων είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό η, τα ε, ε, από τη φύση τους επιβάλλουν τον ε, νόμο αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να επιβάλλουν και να καλύψουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να υπάρξουν νέοι κανόνες που θα λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπασέσκου. Ο κύριος Σέμετο, επίτροπος, έχει το λόγο έτσι ώστε να δώσει την τελική του άποψη όσον αφορά την ε, συζήτηση αυτή. Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι σαφές ότι η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών και η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι κοινή προτεραιότητα για όλους μας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναζητεί να εξεύρει την σωστή ισορροπία με την ενίσχυση της προστασίας πνευματικών ε, δικαιωμάτων και τη διευκόλυνση του παγκοσμίου εμπορίου. Και βλέπουμε και χαιρόμαστε για το ότι συμμερίζονται αυτούς τους στόχους οι ευρωβουλευτές. Επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και ένα ευρύτερο πλαίσιο γεγονότων και στοιχείων σε σχέση με τη διεθνή συνεργασία και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα γενώσιμα φάρμακα διαμετακόμιση ήταν ένα ακαθόδες ζήτημα. Πιστεύω ότι με πολύ προσεκτικό τρόπο το εξετάσαμε παρόλα αυτά και θεσπίσαμε ένα αξιόπιστο πλαίσιο δράσης ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Πολλοί από εσά αναφέρθηκαν σε αυτό το ζήτημα σήμερα και θέλω να σας αναφέρω ότι πρόσφατα γεγονότα σε σχέση με την Ινδία και από πλευράς ε, Υπουργού, Ινδού Υπουργού που ανέφερε τη σπουδαιότητα αυτού του θέματος για τα γενώσιμα φάρμακα που δεν θα ε, δημιουργούν πλέον πρόβλημα στο μέλλον εφ' εξής. Κινούμαστε βλέπω νομίζω στη σωστή κατεύθυνση και σε σχέση με τη διατύπωση που υιοθετήθηκε στην πρότασή μας νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σωστή και λεπτή ισορροπία. Λαμβάνω υπόψη ε, επίσης τις παρατηρήσεις σας σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο σε σχέση με τους ε, τελωνιακούς ε, ή και την ενημέρωση και πληροφόρηση των καταναλωτών δεν υπάρχει κάθε πτυχή σε αυτόν τον κανονισμό. Όμως ε, με τις παρεμβάσεις σας ε, γίνονται ε, χρήσιμες προτάσεις για το πολιετές πρόγραμμα δράσης που πρόκειται να προτείνουμε προσιοθέτηση. Και σε σχέση με τις αλλαγές όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο νομοθεσίας θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με την αναθεώρηση των σημάτων και των τεχνικών στοιχείων ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων προϊόντων. Θα υπάρξει λοιπόν ενημέρωση και το θέμα της διεύρυνσης ε, του πεδίου εφαρμογής. Ε, φυσικά συμφωνούμε ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα περίπλοκο και σύνθετο ζήτημα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό προτείναμε να έχουμε ξεχωριστές διαδικασίες και θα προτείνουμε για τα ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας να υπάρξουν νομικές διαδικασίες που θα καθορίζουν την παραβίαση ε, δικαιωμάτων μέσω των ε, προϊόντων απομίμησης ή πειρατείας και τα τελωνία, οι τελωνιακές αρχές ε, νομίζω είναι ο θετικός, ε, ε, το θετικό επίκεντρο μέσω του οποίου μπορούμε να δράσουμε για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων, συγγενών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να βρούμε απαντήσεις όμως για όλα τα ερωτήματα τα οποία αναφύονται σήμερα. Μόνο ισορροπημένες λύσεις είναι εκείνες που χρειάζονται και πρέπει να εξευρεθούν γοργά ώστε μέχρι τα τέλη του έτους κατά την, τον εορτασμό της 20ης επαιτίου της ενιαίας εσωτερικής αγοράς να έχουμε προχωρήσει. Σας διασφαλίζω ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει και να διευκολύνει αυτές τις διεργασίες. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε Σέμετα. Και τώρα στη συνέχεια ο εισηγητής μας ο κύριος Κρόισμαν θα λάβει τον λόγο και πάλι και καταδεικνύεται και ευχαριστώ για τις συζητήσεις και είναι σαφές ότι οι τελωνιακές αρχές δεν μπορούν να είναι ο διαιτητής όσον αφορά δικαιώματα, ε, ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Πιστεύω ότι οι ανησυχίες που ακούγονται είναι αδικαιολόγητες διότι το κείμενο για τα γενώσιμα διασφαλίζει ότι οι ε, τελωνιακοί υπάλληλοι το την ελεύθερη ελεύθερη διακίνηση ε, γενοσύμων φαρμάκων δεν δικαιούνται να την παρακολύουν. Και σε σχέση με ένα ε, στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε ότι το, οι αρχές του κράτους δικαίου θα πρέπει να διασφαλίζονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκείνος ο οποίος έχει τρωθεί θα, μπορεί να, θα πρέπει να μπορεί να εκφράσει τις ε, επιφυλάξεις του και τις ε, απόψεις του όσον αφορά τα μέτρα τα οποία υιοθετούνται και ιδιαίτερα όσον αφορά το θέμα delegated acts την κατεκπροσώπηση ε, εντολή και δραστηριοποίηση όταν έχουμε μικρές αποστολές που αποτελούνται από τρία το πολύ κομμάτια μέσα σε ένα συγκεκριμένο βάρος. Ελπίζω ότι αύριο στην ψηφοφορία θα υπάρξει ευρύτατη πλειοψηφία ώστε άμεσα να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με τις διαβουλεύσεις ε, με το Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος κατά τα τέλη του έτους να έχουμε επιτέλους ένα κανονισμό που θα αρχίσει να ισχύει, που θα είναι επωφελής υπέρ των δικαιωμάτων των καταναλωτών, υπέρ των επιχειρήσεων, υπέρ όλων εκείνων όπως το τονίστηκε που χρειάζονται αυτή την προστασία και αρρωγή. Και από πλευρά των ε, τελωνιακών αρχών πρέπει να μειωθεί το γραφειοκρατικό βάρος, να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Νομίζω τα καταφέραμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε ως εισηγητής κύριε Κρόισμαν. Έχω θετική εντύπωση που αποκόμισα και έτσι μπορώ να πω ότι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση. Φαίνεται ότι τα ηθικά προβλήματα μπορούν να ε, προκαλέσουν και να συνεπάγονται και οικονομική απώλεια.